αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε και τις σωστές ε, αποφάσεις ε, και να ε, δεσμευτούμε να κάνουμε αυτά που κάναμε πριν να φύγουμε για τις διακοπές, δηλαδή αυτή η Επιτροπή Μεταφορών να καταλήξει σε πραγματικές προτάσεις και η εργατική αυτή μας μέθοδος αλλά και η αγαστή συνεργασία μεταξύ μας να συνεχιστεί. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά ζητήματα θα μας απασχολήσουν και είμαι πολύ ευτυχής που σας ξαναβλέπω. Όλοι είστε μαυρισμένοι, όμορφοι και θα ξεκινήσουμε αυτό το πρώτο σημείο με ψηφοφορίες. Un petit ordre du jour, excusez-moi. Un petit point à l'ordre du jour. Ένα σημείο έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Να σας πω ότι το 6 έχει αναβληθεί και αυτό το σημείο θα συζητηθεί λεπτομερώς στη συνεδρίαση των συντονιστών. Και ξεκινάμε βεβαίως με τις ψηφοφορίες. Θα κάνουμε ένα, μια δοκιμή για να δούμε αν έχετε όλες τις κάρτες σας. Non, mais ça, on le fera après le vote. Ψηφίζουμε λοιπόν να ελέγξουμε τα μηχανήματα και τις κάρτες. Δεν υπάρχει μετάφραση στα Ιταλικά. Πού είναι τα Ιταλικά? Il manque des traductions. Dans cette salle, nous avons un régime limité, hein. mais nous n'avons pas toutes les langues aujourd'hui. Alors, dans les traducteurs, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent... Η πρόεδρος απευθύνεται στους ερμηνείς. Εάν υπάρχει κάποιος που να κάνει γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ρωτάει. Όχι, μου λένε από τους Γερμανούς, από τους Άγγλους, ούτε, όχι, ούτε ούτε. Δεν έχουν προβλεφθεί τα Ιταλικά σήμερα. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε περιορισμένο, περιορισμένη σύνθεση διερμηνής. Όχι, δεν έχουμε ούτε ε, λουξεμβουργικά σήμερα. Donc, nous n'avons pas la traduction italienne. Bon. Où sont nos collègues italiens? Où είναι οι Ιταλοί συνάδελφοί μας? On va essayer. Θα προσπαθήσουμε. Λυπούμε είναι ένα πρόβλημα αίθουσα. και έχουμε μόνο τις γλώσσες των συντονιστών και των αντιπροέδρων προβλέψει για αυτή την αίθουσα όπου δεν χωράνε παραπάνω καμπίνες, παραπάνω γλώσσες. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα λέω αργά για να μην ε, χάσετε τη ψηφοφορίες και ελπίζω πως στο μέλλον δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Alors, au niveau... Πέρα της, ε, της λοιπόν τώρα, έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε με την ψηφοφορία για τον προπολογισμό του 2018. Έκθεσή σας είναι αυτή κύριε Τοζενόφσκι. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα νούμερα των τροπολογιών. Αυτά θα σας λέω, τα νούμερα των τροπολογιών. Τροπολογία 5587. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5750. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5551. Υπέρ, κατά αποχές θα <clears throat> κάνουμε έλεγχο γιατί δεν, δεν ήταν ξεκάθαρο 55-51 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Le vote Τέλος. Απορρίπτεται. 55-52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Τώρα έχουμε τη 5553 και τη 5705. Τις ψηφίζουμε από κοινού υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. Δύο επόμενες τροπολογίες, 5554 και 5706 από κοινού Ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 55-55 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Α, όχι. Εγκρίνεται. C'est la rentrée pour tout le monde. Ναι, και για μας είναι επιστροφή στα θρανία, οπότε... Δύο τώρα ταυτόσημες, 55, 56 και 55, 57. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Amendement 55-80. Qui est pour? 55-80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνονται 5581 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες τώρα, 5558 και 5559 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 5582. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός θέλετε να γίνει. Ωραία. Ψηφίζουμε για την 5582. Πέρασε. Έχετε δίκιο, κύριε Βίμ Βαντεκάμπ. Απορρίπτεται. Τι όπως πάντα, τι λέτε. Ne commençons pas l'année comme ça. Α, όχι, να μην ξεκινήσουμε έτσι τη χρονιά. Συνεχίζουμε τώρα. Τροπολογία 5561. Ίδια με την 5591. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα, ταυτόσημες επίσης 5563, 5578. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 5564 και 5579 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5590 υπέρ κατά εποχές δεν κατάλαβα ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά Le vote est fermé. Τέλος ψηφοφορίας. Η 5590 της Προέδρου εγκρίνεται. 5589 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5570 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55-65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 55-66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55-67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55-68 υπέρ κατά υπέρ κατά να επαληθέσουμε αρχίζει η ψηφοφορία Καλημέρα σας κύριε Κούν πως είστε καλά Εγκρίνεται 55-69. Ποιοι είναι υπέρ. Qui est contre. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55-71. Υπέρ. Α, είναι μαζί με την 55-72, ε, γιατί είναι ταυτόσημες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ακόμα δύο. 55, 73, 55, Ποιοι είναι υπέρ. Αποχές. Εγκρίνονται. Άλλες δύο ταυτόσημες, οι επόμενες δύο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Δύο ταυτόσημες, οι 55-76 και 55-77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5584 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5585 και υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές η 16 εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ Α, 18 συγγνώμη διορθώνει η πρόεδρος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ Υπέρ της 20 ποιος είναι Ναι αλλά προσπαθώ περιμένω μπασκέ Βάρα. Κατά 21 Ποιοι είναι υπέρ Κατά Αποχές Εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Όχι, ήταν ε, σαφές, κυρία Γκραπίνη. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 28 εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές 30 εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές 32 εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές συμβιβαστική 4 εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές η 44 εγκρίνεται 42 υπέρ κατά κα, αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές 53 ε, ε, εγκρίνεται η 59 υπέρ κατά αποχές 59 εγκρίνεται τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 55. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα αυτής της τροπολογίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγινεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ κατά αποχές έγινε, τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές έγινε. τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές έγινε 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η 66 α θέλω έλεγχο ηλεκτρονικό για την 65 Τέλος της Εγκρίνεται. 65 λοιπόν εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου και αυτό ηλεκτρονικά. Je ferme le Τέλος ψηφοφορίας. Συν 39. Μείον μία. Εγκρίνεται. Λοιπόν, μπράβο στον εισηγητή. Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε λοιπόν.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

Allons-y, nous reprenons nos travaux. Je rappelle que le point 6 à l'ordre du jour a été reporté. Ξαναρχίζουμε. Σας θυμίζω ότι το 6 έχει αναβληθεί. Και έχουμε τώρα την παροπισίαση. μάλλον θα προχωρήσουμε με την προ... το σημείο 5 την προώθηση της χρήσης της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την οδηγία του 2009 για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένας από τους τομείς ε, ε, ε, δράσεων κλειδιών Γι' αυτό το είναι θέμα προτεραιότητας και γι' αυτό και εμείς θα υποβάλουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ήτρε. Έχουμε λάβει περίπου 200 τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης, αλλά ο εισηγητής μας, ο κ. Βάσ Έκχαουτ, θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο, γιατί ήδη έχει γίνει ανταλλαγή απόψεων από αυτού. Κύριε Βίμ, Βαντεκάμ και κύριε Βικτόρ, μπορείτε να μιλάτε πιο σιγά για να μην ενοχλείτε τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Βίμ Βαντεκάμ πάντα μας δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Οι Ολλανδοί δεν είναι ποτέ ε, ήσυχοι. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ασχοληθούμε με τις τροπολογίες 222 έχουμε, όπως είπατε. Σχετικά μικρός ε, αριθμό, Μας έχουν συμβεί και χειρότερα. Μη σας εκπλήσει. Γνωμοδότηση είναι, ναι. Αλλά είμαι και στην ένβη εισηγητή, όπου έχουμε 1111. Δηλαδή εκεί έχουμε τέσσερι άσου στη σειρά και εδώ έχουμε τρία διάρκεια στη σειρά, για να θυμάστε τον αριθμό των τροπολογιών. Αν δείτε τις τροπολογίες, θα δείτε ότι αφορούν πολλά και διαφορετικά ζητήματα και θα αποτελέσει για μας μια πρόκληση να βρούμε τη σωστή συμβιβαστική λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια συνεδρίαση και στο Στρασβούργο θα ακολουθήσει άλλη μια συνεδρίαση και αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος μετά. Προσπαθούμε να δούμε μήπως τυχόν μπορούμε να το παρατείνουμε λίγο για να έχουμε και μια τρίτη συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα χρειαστεί. Αυτό που θα ήθελα για την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών την επόμενη εβδομάδα είναι να γίνει μια συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές για να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Δεν θα δώσω δηλαδή εγώ τις δικές μου προτάσεις απευθείας, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ διαφοροποιημένο το πλαίσιο. Θέλω πρώτα να ακούσω τις προτεραιότητες των σχεδόν εισηγητών. Και βεβαίως θα μου ήταν πολύ χρήσιμο αν θα μπορούσε τώρα όποιο έχει κάποια ζητήματα να αναφέρει στην ανταλλαγή απόψεων. Προτιμούν βέβαια οι σκιώδει σύγητε να το κάνουν σε μια πιο περιορισμένη σύνθεση μόνο με σκιώδει σύγητε. Πάντω είναι πολύ σημαντικό αυτό θέλουμε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη συναντήση με του σκιώδει σύγητε και μετά να δούμε προ ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε για τι συμβιβαστικέ λύσει. Πολύ σύντομα θέλω να σα πω αυτά τα οποία έχω κατά νου. Πρώτον, πρέπει να δούμε αν θα χρειαστούμε χωριστό στόχο για τον τομέα των μεταφορών. Ορισμένε τροπολογίε αυτό προσπαθούν να κάνουν θα έχουμε και κάποια ανώτατα όρια για προηγμένα καύσιμα, για επόμενη γενιά καύσιμα κλπ. κλπ. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό. Θέλουμε να έχουμε ένα συνολικό στόχο των μεταφορών χωρίς ε, να το επιβαρύνουμε με πάρα πολλούς επιμέρους στόχους. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε με τους χειώδεις εισηγητές. Κάποιο ανώτατο όριο για τα βιοκαύσιμα ε, αρκετά ζητήματα που συνδέονται και με τα θέματα της, των κριτηρίων βιωσιμότητας. Όσο πιο ισχυροί είμαστε για τα κριτήρια βιωσιμότητας, τόσο περισσότερο φαντάζομαι ότι θα πούν κάποιοι σκιώδεις συγητές ότι δεν χρειαζόμαστε ανώτατο όριο ή μπορούμε να έχουμε χαμηλότερο, χαμηλότερο ανώτατο όριο. Όπως σας είπα, θέλω να ακούσω τη γνώμη των σκιωδών εισηγητών. Και έχουμε και μια νέα κατηγορία όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, τα βιώσιμα και τα υψηλή βιωσιμότητα. Και εδώ πάλι θέλω να ακούσω το σκεπτικό για τέτοιου είδου ε, αλλαγέ. Θα γίνει μια συζήτηση επίσης για το παράρτημα 9. Κάποιοι τροποποιούν το παράρτημα 9 και συμφωνώ γιατί ξέρουμε ότι κάποια από αυτά, όπως οι μελάσσε κλπ, χρησιμοποιούνται και για βιομηχανικές πρακτικές και υπάρχει ο κίνδυνος ότι αν μπουν στα προηγμένα βιοκαύσιμα θα υπάρχουν αποτελέσματα μετατόπισης σε βιομηχανικό επίπεδο στη βιομηχανία τροφίμων και στη χημική βιομηχανία. Είναι ένα θέμα λοιπόν που έχει επισημανθεί και πρέπει να το συζητήσουμε. Ακόμη, κάποιες τροπολογίες βάζουν ε, μηδέν όριο, δηλαδή ε, απαγορεύουν ε, τα ενεργειακά φυτά. Ξέρω τη συζήτηση για το φινικέλαιο, αλλά αν απαγορεύσουμε συγκεκριμένα προϊόντα θα μπούμε σε διεθνεί συζητήσει από αυτόν. Θα προτιμούσα λοιπόν να έχουμε ισχυρότερα κριτήρια, τα οποία θα ισχύουν για όλους και βέβαια θα γνωρίζουμε ότι το φινικέλαιο θα έχει περισσότερες δυσκολίες στο να πληρεί τα κριτήρια αυτά παρά να απαγορεύσουμε κάποια συγκεκριμένα ενεργειακά φυτά. Αυτό θα μας δημιουργούσε προβλήματα. Άλλο ένα θέμα λοιπόν που θέλω να συζητήσω με τους χειώδεις συζητητές. Αυτά λοιπόν και την επόμενη εβδομάδα προσβλέπω στις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Έρχεται η συζήτηση. Και δίνω το λόγο στον κύριο Σαλίνη. Μπορείτε να μιλήσετε ιταλικά γιατί θα σας μεταφράσουν ε, για μας. Ε, Ναι. Η θέση του ΕΛΚΕ για την έκθεση αυτή είναι αρκετά σαφής και συνάδει και με τη θέση που τηρούμε για το ίδιο θέμα και στις άλλες επιτροπές, ε, κυρίως στην Ήτρη και στην ΕΜΠΗ. Θα σταθώ λοιπόν πολύ σύντομα σε τρία πράγματα, τρία άρθρα, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για την Επιτροπή Μεταφορών. Για το άρθρο 3, ο στόχος του 27% ή του 35% ή του 45% ανάλογα με την πολιτική ομάδα, ε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τον συζητήσουμε. Ο δικός μας ο στόχος ε, είναι ένα 27% γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ο σωστός στόχος για να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειων και ενέργειας και των άλλων πηγών που ε, αφορούν το μέλλον της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρώπης. Ε, τώρα, στο ίδιο κεφάλαιο πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο συμβιβασμό για τον προηγούμενο στόχο του 10% που αφορά τις μεταφορές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση για το θέμα αυτό και φυσικά ε, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να παραμείνει αυτός ο στόχος του 10% όπως είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει επικοδομητική συζήτηση από αυτού με τον εισηγητή. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 7, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει σχέση και με το άρθρο 25. Στο άρθρο 7 υπάρχει ε, ισχυρή αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή, ε, βάσει της οποίας ε, σωστά πρέπει η Επιτροπή Μεταφορών να, να εκφράζει τακτικά τις προτεραιότητές της. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 7 και έχουμε και το θέμα της μετάβασης ε, των βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς ε, και την αλλαγή τους με βιοκαύσιμα ε, δεύτερης γενιάς. Εδώ έχουμε προτείνει ε, το ανώτατο όριο του 7% να μείνει μέχρι το 2030, ώστε η μετάβαση στην οποία πιστεύουμε να γίνει ε, λογικά και βαθμιδών χωρίς να διακυβευτεί και η σχέση εμπιστοσύνη που έχουμε δημιουργήσει με του Ευρωπαίου επενδυτέ όταν του προτείναμε να επενδύσουν σε βιοκαύσιμα πρώτη γενεά. Σωστά να γίνει η μετάβαση, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε η Ευρώπη να μην χάσει επενδυτέ. Το άρθρο 25 ε, αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα. Εγώ θα σταθώ στο πρόβλημα το οποίο μόλις υπενθύμησε και ο εισηγητής του παρατήματος 9. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να διευρύνουμε τα όρια, να μην είναι ευέλικτο δηλαδή το παράρτημα 9. Όπως ε, ακούστηκε οι ζωοτροφές, δηλαδή προϊόντα τα οποία αναφέρονται αυτή τη στιγμή στο παράρτημα 9, χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις, ε, υπήρχε για παράδειγμα η περίπτωση της μελάσας ε, και σε άλλες ε, παραγωγικές αλυσίδες. Το παράρτημα 9 λοιπόν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο απόβλητα και όχι σύνθετα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται και αλλού. Ε, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουμε σχέση με άλλες γραμμές παραγωγής. Ε, ε, και το θέμα αφορά και τη χημική βιομηχανία, αλλά όχι μόνον αυτή. Και πιστεύω ότι προς τιμήν και ενό εκ των πυλώνων της κυκλικής οικονομίας, ένα προϊόν όταν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο, θεωρούμε ότι είναι άχρηστο να χρησιμοποιείται και πάλι εντός αυτής της κατηγορίας, που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετάβαση από την ε, από τα βιοκαύσιμα πρώτης γενεάς στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Αυτές λοιπόν είναι οι θέσεις μας. Ε, είμαι καθόλου διατεθειμένος να συνεργαστώ με τον εισηγητή όπως κάναμε και μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ε, καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Για το θέμα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε χρήσιμες συνεδριάσεις των σκιωδών εισηγητών, διότι πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ευρύ, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό και ενώπιον των άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα ε, εύρωστο κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία. Διαπιστώνω ότι υπάρχει συνένεση ως προς τη διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ των διαφόρων ε, βιοκαυσίμων ε, γιατί δεν έχουν όλα την ίδια ισότητα και φυσικά δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε διατροφικές κρίσεις και να επιδεινώσουμε την αποψήλωση που έχουν θέματα τα οποία έχουν συνέπειες και στην κλιματική αλλαγή. Βέβαια, το ποια θα πρέπει να είναι αυτά τα προϊόντα πρέπει ακόμα να τα συζητήσουμε. Εμεί ω σοσιαλδημοκράτε πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και το κόστο των φυτών που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο παραγωγή, αλλά και τον τρόπο ε, αλλαγή τη χρήση των γεών, το, παρα, το περιβόητο iLook. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ χρησιμοποιούνται τα καύσιμα ε, νομίζω ότι αυτό είπε και ο εισηγητή και οι σκιώδεις εισηγητές και θα πρέπει να εμβαθύνουμε τη συζήτηση αυτή για να έχουμε μια συνένεση στα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα των εκπομπών, αλλά δεν είναι τα μόνα που πρέπει να συνυπολογίσουμε στους υπολογισμού μας αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικά στοιχεία. Ε, πρέπει να συζητήσουμε καλύτερα επίσης και τα ποσοστά, αυτό το είπαμε, τα ανώτατα όρια των βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς, ε, ε, τα όρια των ε, προϊόντων που προωθούνται και επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν και εθνικοί στόχοι πέραν των ευρωπαϊκών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς συμφωνούμε με αυτή την ιδέα και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει στις διαπραγματεύσεις με μια ισχυρή και ενωμένη θέση, κυρίως για το άρθρο 25 με το Συμβούλιο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε και πιο ήπια θέση για τα συνολικά όρια, για παράδειγμα 9% του 6,8% αλλά με πιο περιορισμένο ορισμό των καθαρών βιοκαυσίμων και να λαμβάνουμε υπόψη και τα στοιχεία του ILOC. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα προηγούμενα ε, ε, βιοκαύσιμα 5,3% σε σχέση με το 3,5% που είχαμε το 2005 και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την ηγεμονία των ορυκτών καυσίμων. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι ε, εάν λάβουμε υπόψη τους πολλοπλασιαστικούς παράγοντες, δηλαδή το γεγονός ότι υπολογίζουμε 2, 3 ή τέσσερις φορές παραπάνω κάποια καύσιμα για να δώσουμε μεγαλύτερη δυνατότητα σε κάποιους τομείς, για παράδειγμα στην αεροπορία, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε καθαρές ενέργειες και δεν θα πρέπει να δημιουργείται χάσμα στην νομοθεσία και να δημιουργούνται στρεβλώσεις ε, ε, για να μην χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα. Ε, περιμένω λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε στις συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών για να καταλήξουμε σε, σε περάσματα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντέμες Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που συνεισέφεραν στη συζήτηση. Από τις τροπολογίες ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ε, γνωμοδότηση και για την Επιτροπή μας αλλά και για το Κοινοβούλιο εν γέννη. Με χαρά διαπιστώνω ότι μία σειρά από τις τροπολογίες μας ε, υποστηρίζονται και από άλλες πολιτικές ομάδες, η κυκλική οικονομία, η αλυσίδα της βιομάζας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία στα οποία βέβαια διαφέρει η απόψή μας από τη θέση του εισηγητή, αλλά αυτό είναι λογικό. Ήθελα να πω ότι κάποιες ομάδες ζητούν να υπάρχουν δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι, όπως αυτούς που γνωρίζουμε. Για μας, ε, δεσμευτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χωρίς ε, να υπάρχει και δεσμευτικός στόχος σε εθνικό επίπεδο, θα ήταν πιο αποτελεσματικό, φθηνότερο και προσφέρει και τις ίδιες εγγυήσεις για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας σε διεθνές επίπεδο, που είναι αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι. Επιπλέον διαπιστώνω ότι κάποιοι ζητούν να αυξηθούν τα ποσοστά των ευρωπαϊκών στόχων, να πάμε από το 27% στο 30% και κάποιοι φτάνουν και μέχρι και το 35%. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ευρωπαϊκός στόχος να είναι ρεαλιστικός, να μπορεί να επιτευχθεί και να μην ε, ε, είναι ει βάρο της ανταγωνιστικότητάς μας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ε, δραματικό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να υπάρχει συνένεση αφενός και ρεαλισμός αφετέρου. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ του 27% στόχος, όπως συμφωνήθηκε και στο Συμβούλιο άλλωστε. Γνωρίζουμε ότι τα βιοκάψιμα πρώτης γενεάς πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται σιγά σιγά. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με έξυπνο λογικό τρόπο ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες και να αποφύγουμε και την έλλειψη ασφάλειας για τους επενδυτές. Ιδάλλως θα χάσουμε την υποστήριξη για τα πιο προηγμένα βιοκαύσιμα. η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μείωση της τάξης του 20% μέχρι το 2020. Είναι κοντά στο στόχο αυτό. Είναι καλή η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίξουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντέμες Μάκερ. Ο κύριος Ραντός έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την, ε, την παρουσίαση αυτού του θέματος ε, για τη μείωση των καυσίμων πρώτης γενιάς από 7% στα 3,8%. Όμως, δεν είναι σαφές πώς θα επιτύχουμε το στόχο αυτό. πώς θα ανανεώσουν τα ανανεώσιμα δεύτερης γενιάς, τα ανανεώσιμα πρώτης γενιάς. Οι περισσότερες τροπολογίες και οι δικοί μου μαζί προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, δηλαδή να κρατήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων καυσίμων πρώτης γενιάς. Δεν ξέρουμε πώς θα επιτύχουμε το στόχο του 3,8% για τα κάψιμα δεύτερης ε, γενιάς. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε το στόχο ε, της μείωσης των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα, να έχουμε ενεργειακή αποτελεσματικότητα και να μην καταργήσουμε τις προσπάθειες για τα καύσιμα πρώτης γενιάς. Αυτή θα είναι η γραμμή των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, η κυρία Άντερσον. Καλημέρα συμφωνώ με τους στόχους ε, αυτού του κειμένου και είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρούς στόχους, ό,τι και αν προκύψει τελικά. Θέλω να επισημάνω το άρθρο 2. Χρειαζόμαστε ε, έναν ορισμό της τομεακής ολοκλήρωσης σε αυτό το τομέα, γιατί είναι εύκολο να λέμε αυτά που λέμε, αλλά αν δεν δώσουμε ορισμούς στα ευρωπαϊκά νομιμοθετικά κείμενα και αν δεν τονίσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός και το υδρογόνο θα έχουμε δυσκολίες. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα οποία κάνουμε εδώ θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των συνολικών υποχρεώσεών μας βάσει της συνθήκης, να προωθήσουμε δηλαδή την περιβαλλοντική προστασία οποτεδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Ελπίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα μπορέσει να εκφράσει μια ισχυρή θέση και ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστούμε κυρία Άντεσον, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα συμφωνήσω με την ανάγκη να προχωρήσει αυτή η αναθεώρηση και η αύξηση των στόχων. Επειδή όταν είχαμε την έκθεση Τούρμες ε, ήμουνα η πρώτη συντάκτρια γνωμοδότησης ε, από πλευράς Επιτροπής Μεταφορών και τότε έγινε η όλη συζήτηση για τη δαιμονοποίηση ε, η οποία ξεκίνησε από καλή διάθεση του κυρίου Άικχουτ, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν συζητάμε για ενέργεια βρισκόμαστε ενώπιον μιας βάναυσης ε, μάχης ε, για τα διάφορα συμφέροντα και θα πρέπει να τα δούμε αυτά. Προσπαθούμε ε, να μην βάλουμε αυτά που δεν θέλουμε στο χρονοδιάγραμμα, γιατί παρόλο το γεγονός ότι ξεκινά από καλή διάθεση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην δαιμονοποιήσουμε τα βιοκαύσιμα από την αρχή, διότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ε, προς τα που κατευθύνεται η ΚΑΠ και πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε αρκετά θέματα, να μην τα συνδέσουμε τόσο πολύ με το θέμα της αποψήλωσης των δασών, αλλά ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Υπάρχει και το θέμα της κυκλικής οικονομίας, το οποίο δεν θα πρέπει εδώ να λησμονούμε. Θα πρέπει να δούμε πώς συνεισφέρει η βιομάζα στις μεταφορές και θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν αρκεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε ή αν θα έπρεπε να επιταχύνουμε. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αϊκούτ αν μπορούμε να προσθέσουμε και κάτι το οποίο να αφορά ε, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθεί στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αφενό ε, να μην υπάρχουν ε, ε, χρηματοοικονομικά μέσα και κίνητρα για την εφαρμογή των οδικών δικτύων στα νέα αιτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων και εδώ υπάρχει και μια αντιπαράθεση και είναι και λίγο παράδοξο αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τον τομέα της αεροπορίας και της ναυτιλίας, θα ήθελε να είναι λίγο πιο σαφή αυτά τα οποία μας είπε. Ε, να μην τους θεωρούμε απλώς έναν ακόμα κλάδο λαμβάνοντας υπόψη τι θα μπορούσαν να κάνουν, αλλά να δούμε και ε, πώς μπορούν να συνεισφέρουν διαφορετικά. Ε, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γιάννα Σέντερ. Κύριος Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να απαντήσω στο σχόλιο του εισηγητού για το αν πρέπει να έχουμε κριτήρια ή κάποια απαγόρευση για συγκεκριμένα προϊόντα. Συμφωνώ απολύτως με την ιδέα του να έχουμε ισχυρά και σαφή κριτήρια τα οποία θα μας καθοδηγούν προς λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να έχουμε περιπτώσεις όπου ε, είχαμε απαγορεύσεις ή επιδοτήσαμε ένα προϊόν και απαγορεύτηκε κάποιο άλλο και τελικά δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Νομίζω ότι τα ισχυρά κριτήρια είναι σημαντικά και η αγορά θα μπορέσει να επιλύσει αυτά τα θέματα με βάση τα κριτήρια. Τα λέω όλα αυτά γιατί εγώ είμαι από τη Βόρεια Σουηδία όπου έχουμε τεράστια δάση, ίσως τα έχετε δει, ίσως τα έχετε επισκεφθεί. Την ξυλία τη χρησιμοποιούμε είτε για κατασκευή οικειών είτε ως καύσιμο και επί εκατοντάδες χρόνια το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τα δάση όλοι γνωρίζουν ότι είναι θετικά για το περιβάλλον. Το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες λύσεις. Και στη Βόρεια Ευρώπη τα δάση είναι ένας πόρος που μπορεί να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νίλσεν. Και στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω το λόγο στον κύριο Βόλπη από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνεδρίασή μας κύριε Βόλπη. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις για τα θέματα που αναφέρθηκαν και να μας μιλήσετε και για τη στρατηγική και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτές για τα σχόλιά τους. Είδαμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και έχω πέντε σημαντικά σχόλια. Καταρχήν το στόχο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ξέρουμε ότι κάποιες πολιτικές ομάδες ε, ζητούν να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και δεν μας εκπλήσει γιατί και στο παρελθόν ε, η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ε, υπέρ ενός στόχου 5%. Ε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις της συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Και έχουμε κάποια σχόλια, ιδίω για το ρόλο της βιοενέργειας που καλύπτει το 60% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνοντα προς το 2030 θα συνεχίσει να έχει ένα υψηλό μερίδιο παρότι μειώνεται κατά 50%. Το να έχουμε δύο ειδών κριτήρια βιωσιμότητα, περιορίζοντας τη χρήση των βιοκαυσίμων και της βιομάζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζει την αποδοτικότητα και την ικανότητα να επιτύχουμε ε, το στόχο του 27% και τους στόχους ε, που είναι πιο φιλόδοξοι όπως προτείνονται από κάποια κρατημέλη. Το δεύτερο σχολείο μου αφορά το στόχο για τις μεταφορές. Κάποιες πολιτικές ομάδες και εδώ θέλουν ένα συγκεκριμένο στόχο για τις μεταφορές. Εδώ συμφωνώ με την ερώτηση του εισηγητού για το σκεπτικό σχετικά με αυτό το στόχο για τις μεταφορές. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζονται στο στόχο του να έχουμε μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στα μέτρα που λαμβάνονται. Ε, ε, υπάρχει ο στόχος του τουλάχιστον 27% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κινούμεθα προς εναρμονισμένα μέτρα σε διάφορους τομείς και συγκεκριμένα στον τομέα των μεταφορών έχουμε προτείνει οι προμηθευτές ε, να έχουν μια υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν καθαρά καύσιμα στο πλαίσιο της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει από την εφαρμογή της ε, τωρινής οδηγίας. Έχουμε δει ότι ε, ένας στόχος για τις μεταφορές δίνει μικρότερη διαβελιξία στα κράτη-μέλη και δημιουργεί και κάποια προβλήματα για την διαφοροποιημένη υλοποίηση σε κάθε κράτος μέλος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμεί να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών για να έχουμε μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και εδώ υπάρχει ε, μεγάλη ε, τάση προς την διαφοροποίηση ε, ώστε να αποφύγουμε τα ορυκτά καύσιμα και αυτό το προτιμούμε από το να έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Τέλος, το θέμα της επίπτωσης της έμεσης αλλαγής χρήσεων γης, του ILUC. Κάποιοι ευρωβουλευτές συμφωνούν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή μετάβαση, μετάβαση από τα καύσιμα πρώτης γενιάς στα καύσιμα δεύτερης γενιάς στην υλοποίηση της οδηγίας για τα ανανεώσιμα καύσιμα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ ε, τις ε, ε, παρενέργειες της οδηγίας για τη χρήση γης και η Επιτροπή θα βασιστεί στη συζήτηση αυτή που έχει γίνει, θα επωφεληθεί από τα συμπεράσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ξέρουμε ότι η έμεση αλλαγή χρήσεων γης μπορεί να αποτελέσει ένα ζήτημα, ιδίως για τα βιοκαύσιμα δεύτερη γενιά, αλλά θα είναι προτιμότερο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό μειώνοντα τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων δόδιμων φυτών. Αντί να βάλουμε παράγοντες που αφορούν το iLook στη μεθοδολογία μας, στη μεθοδολογία των αερίων του θερμοκηπίου γιατί αυτό αφορά τις άμεσες εκπομπές. Αν βάλουμε και τις έμεσες εκπομπές όπου υπάρχει αβεβαιότητα, δεν ε, είναι λύση που ταιριάζει με την τωρινή μεθοδολογία. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της έμεσης αλλαγής χρήσεων γης, μειώνοντας τα βιοκαύσιμα ε, βάσει δόδιμων φυτών και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι το μερίδιο αυτών των βιοκαυσίμων θέλουμε να το επαναφέρουμε στα επίπεδα πριν από το 2009. Δηλαδή πριν από την τωρινή οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα μειώσει σημαντικά την επίπτωση του iLook. Θέλουμε να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και των σημαντικών επενδύσεων που έχουν γίνει στον τομέα αυτό και να επιτρέπουμε στους παραγωγούς βιοκαυσίμων και στους αγρότες να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Και ένα σχόλιο για την νέα αυτή έννοια της υψηλής βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα ανησυχούμε λίγο για το σκεπτικό το μοντέλο που έχουμε δείχνει ότι κάποια βιοκαύσιμα βάσει εδόδημων φυτών, ακόμη και αν έχουν λιγότερες εκπομπές από άλλα, δεν είναι χαμηλού κινδύνου και δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποκλείονται από, την, από το ανώτατο όριο ή να συμπεριλαμβάνονται ως προηγμένα καύσιμα στην υποχρέωση ανάμειξης καυσίμων για τους προμηθευτές. Τέλος, για το παράρτημα 9, έθεσαν ε, κάποιοι ευρωβουλευτές το θέμα αυτό και θέλω να πω ότι η δική μας προσέγγιση βασίζεται στην οδηγία του ILUC. Τη διαπραγματευτήκαμε πριν από δύο χρόνια, την εφαρμόζουν κάποια κράτη-μέλη, την λαμβάνει υπόψη ε, ο κλάδος. Εξετάζουμε λοιπόν το παράρτημα 9 και το χρησιμοποιούμε ως βάση για τον ορισμό των προηγμένων βιοκαυσίμων. Ακόμη να σας πω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός στην οδηγία βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια επανεξέταση της αγοράς κάθε δύο χρόνια. Αν κάποια εδόδημα φυτά ε, αφαιρεθούν, δημιουργείται κάποια νομική αβεβαιότητα για τα προηγούμενα καύσιμα και αυτό θα αποτρέψει τους ε, επενδυτές. Θέλω να σας πω ότι ε, οι στόχοι αυτοί δεν θα υπολογίζονται στους στόχους των δύο καυσίμων, αλλά υπάρχουν στην υποχρέωση των προμηθευτών για ανάμεξη καυσίμων γιατί συνεισφέρουν στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και στη διαφοροποίηση που είναι στόχος για τον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Μπάς Εκχάουτ. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις συμβολές σας. Πιστεύω πως ε, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζουμε τα κεντρικά ζητήματα που, όπως προέκυψαν και από αυτή τη συζήτηση, είμαστε πολύ καλοί στον εντοπισμό των θεμάτων. Ε, τώρα να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε και τις συμβιβαστικέ. Αυτό θα είναι κάπως πιο δύσκολο. Γενικά για τους στόχους βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε και θέλω να τονίσω ότι η Επιτροπή Μεταφορών ε, και μάλλον η γνωμοδότηση για το γενικό στόχο για τα ανανεώσιμες δεν θα είναι αυτό που οι περισσότεροι θα δουν. Θα είναι πολλή συζήτηση, η πολύ πολιτική φύση συζήτηση θα καταλήξει στην Ολομέλεια. Ξέρουμε ότι η Ήτρε είναι αρμόδια επί της ουσίας και αυτό που θα είναι σημαντικό θα είναι ο γενικός στόχος και αυτό θα είναι ένας από, τους βασικούς, τα βασικά θέματα που θα κοιτάξει ο κόσμος. Ε, νομίζω όμως πως αυτή τη γνωμοδότηση μπορούμε να, να κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά την ε, νομοθέτηση Έχουμε γενικούς ε, πολιτικού στόχου που θα προσελκύσουν την προσοχή και η δική μα νομοδότηση δεν θα αλλάξει και τον κόσμο. Θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, ελπίζω πως θα αποφύγουμε να μπούμε σε συζήτηση για αυτή την γνωμοδότηση να ήταν το πιο σημαντικό αυτό. Υπάρχουν κάποια θέματα που συνδέονται με τις μεταφορές που είναι πιο σημαντικά για αυτή την Επιτροπή από ότι ο γενικός στόχος. Δεν λέω πως δεν είναι ε, σημαντικός, αλλά ξέρουμε πώς καταλήγουν ορισμένες από τις νομοδοτήσεις. Δεν θα μιλήσω και για τα όσα είπε η Κομισιόν για το γενικό στόχο, γιατί αν αρχίσω να μιλάω θα μιλάω για κάνα μισάωρο. Τώρα, εξετάζοντας τις συμβαστικές, έχω την εντύπωση ότι για τα προηγμένα βιοκαύσιμα έχουμε κάνει πρόεδρο, κάνουμε πρόοδο και το βλέπω από διάφορες πλευρές του Κοινοβουλίου ότι το ζήτημα θα πρέπει να είμαστε μόνο στη βάση του καλύτερου προσδιορισμού του παραρτήματος 9 ότι θα πρέπει να υπάρχει λιγότερο ανταγωνισμό με εφαρμογέ ε, βιομηχανικές ή της ε, βιομηχανία τροφίμων και ότι αυτό είναι πιο θετικό από την άποψη τη οικονομία. Το άκουσα από πολλού και πιστεύω πως μια συμβαστική είναι σημαντική γιατί έτσι έχουμε καλύτερο ορισμό ε, γιατί βλέπουμε τώρα τι σημαίνει προηγμένα βιοκαύσιμα. Αυτά λοιπόν για την πρώτη γενιά, με τη βάση το, επί τη βάση των τροφίμων, εργαζόμαστε για βιώσιμα βιοκαύσιμα από τρόφιμα, με βάση τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει κάποια ασφάλεια για τους επενδυτές. Η λύση λοιπόν θα είναι να δούμε τα κριτήρια, να εξετάσουμε τα κριτήρια. Και αυτό ισχύει και για τα όσα είπε ο κύριος Νίλσον. Καλύτερα, ισχυρότερα κριτήρια και όχι να αρχίσουμε να απαγορεύουμε κάποια προϊόντα πράγμα που κάνουν άλλες ομάδες όπως η Γκουε για παράδειγμα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που λέει η Κομισιόν δεν αρκεί γιατί αυτό που κάνουμε αυτό το ανώτατο όριο είναι ένα πολύ απότομο εργαλείο, πολύ ε, κάθετο, γιατί ναι, βεβαίως, τότε θα μειωθεί η χρήση των καυσίμων, αλλά είναι πολύ απόλυτο, γιατί δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διακρίνουμε καλύτερα ανάμεσα σε όλα αυτά, αν θέλουμε δηλαδή ένα πιο απόλυτο, ένα πιο λεπτό ε, εργαλείο ε, για να, κάνουμε, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με το ανώτατο όριο. Εγώ πιστεύω πως έτσι πρέπει να το προσεγγίσουμε για να δούμε αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε και σε μια καλή συμβιβαστική ε, ξέρω πως η Κομισιόν δεν θα τις πολύ αρέσουν όλα αυτά, αλλά εμείς είμαστε το Κοινοβούλιο και γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόταση θέλουμε την επόμενη εβδομάδα να βγει, γιατί θέλω να συζητήσουμε λεπτομερώς για αυτά τα ζητήματα με τους συναδέλφους, για να μπορέσουμε επί τη βάση όλων αυτών να προτείνουμε πράγματα και να, βγούμε, να βρούμε συμβαστικές όπου θα έχουμε μεγάλη υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Θυμίζω ότι η 12 Οκτωβρίου θα πρέπει να ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση και να θυμίσω και το εξής την ε, φάση των μεγάλων, ε, των σπουδαίων ε, λόγων και ομιλιών είδαμε στην, την COP21. Είμαστε στην παραμονή της COP23 και η Ευρώπη πρέπει να ξαναπάρει την ηγεσία, την πρωτοπορία σε αυτά τα θέματα για την προοπτική των ε, νέων πηγών ενέργειας. Ελπίζω όντως πως αυτή η έκθεση θα είναι φιλόδοξη. Προχωρήσαμε ε, Τώρα έχουμε φέρει πιο μπροστά το θέμα της ε, παρουσίασης της Κομισιόν για την εφαρμογή του ΕΤΤ. Κύριε Ρότερς, μη φοβάστε, ελάτε εδώ δίπλα μου. Α, δεν θέλετε να έρθετε δίπλα μου, Είστε πολύ συνετός και φρόνιμος. Μπράβο. Α, θα έρθετε τελικά. Ça va Et toi Alors, Ε, δεν χρειάζεται πλέον να σας το συστήσω τον ε, ε, διευθυντή της DG Move. Θα μας ε, κάνετε λοιπόν αυτή τη σύντομη παρουσίαση γιατί 2014 με 2015. Merci, Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι μετά από τις διακοπές. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε χρόνο για να σας παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση για την εφαρμογή των δικτύων RT των διευρωπαϊκών δικτύων για το 2014-2015. Θα περάσω στα αγγλικά τώρα γιατί η παρουσίαση είναι στα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη. Κυρίες και κύριοι, με χαρά σας παρουσιάζω την έκθεση πρόοδου για την εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων 2014-2015 ε, και να σας πω γιατί είμαστε εδώ. Ο κανονισμός προβλέπει να γίνεται μία έκθεση κάθε δύο χρόνια προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω το άρθρο, αλλά απλώς ε, σας υπενθυμίζουμε ότι ε, επ' αυτής της βάσης γίνονται όλα. Πρέπει κάθε δύο χρόνια να σας υποβάλουμε μια έκθεση. Αυτά λοιπόν τα οποία θα σας ε, λέμε ε, είναι πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων και υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν για τα διάφορα μέσα μεταφορών. Τα βλέπετε αυτά στην επόμενη διαφάνεια, όπου διαπιστώνεται ότι σιγά σιγά προχωρούμε και εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια. Για παράδειγμα για τους σιδηροδρόμους και την ηλεκτροδότησή τους, ε, ε διάφορα θέματα που γίνονται στην αυτιλία. Υπάρχουν κάποια ποσοστά επιτυχίας. Ε, η ημερομηνία βέβαια για το βασικό δίκτυο είναι 2030 και η τελική καταληκτική ημερομηνία είναι 2050. Είμαστε πάνω από το ε, 75% σε κάποια πράγματα, σε κάποια είμαστε πιο κάτω, τα παρουσιάζουμε για να ξέρετε πού ακριβώ βρισκόμαστε. Πιστεύουμε ότι προχωρούμε καλά και σας δείχνουμε και στην επόμενη διαφάνεια που βρισκόμαστε και ως προς την οικονομική εφαρμογή και εδώ στη διαφάνεια βλέπετε με μπλε τις δαπάνε που έγιναν και φυσικά με κόκκινο και τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων που είχαμε. Και εδώ θα πρέπει να σας εξηγήσω λίγο τη διαφορά. Βλέπετε ότι στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στο Connecting Europe Facility ότι είχαμε περίπου χαμηλές πληρωμές και υψηλές δεσμεύσεις, ενώ ε, στα ε, ταμεία του ε, τα τα ταμεία είχαμε υψηλότερες πληρωμές και χαμηλότερες δεσμεύσεις. Αυτό είναι λογικό, διότι ξέρετε ότι στην αρχή είχαμε πολύ αυξημένη εφαρμογή όλων των ε, ε, θεμάτων του Connecting Europe ε, Facility και τα πρώτα δύο χρόνια είχαμε μεγάλες δεσμεύσεις κονδυλίων. Ήμουν εδώ, άλλωστε θα θυμάστε πριν από τις διακοπές, για να σας επενθυμίσω τι ακριβώ έγινε με την τρίτη πρόσκληση υποβολή ε, προσφορών και εκεί ήμασταν πάνω από το 95% όταν συμπεριλάβαμε και αυτά. Μας, μας απομένει λοιπόν μόνο ένα 5% του προπολογισμού. Σημαίνει ότι ήταν πολύ ψηλε οι δεσμεύσει το 2014 και 2015, όπως επίσης και για το 2016 και το 2017. Αυτό το βλέπετε στο κόκκινο τμήμα του Connecting Europe Facility. Ε, το μπλε τμήμα είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε στο πρώτο τμήμα της περίοδου και είχαμε και πληρωμές ε, των δράσεων που έρθαν από το προηγούμενο πρόγραμμα των ε, ε διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, στα άλλα ταμεία έχουμε ακριβώς το αντίθετο, γιατί ακόμα είχαμε πληρωμές ε, προγραμμάτων ε, της προγραμματικής περίοδου του 2007-2013 και οι δεσμεύσεις για τις νέες δράσεις ήταν χαμηλότερες από την άλλη πλευρά. Αυτό όμως είναι λογικά, θα το δείτε στο τέλος της περίοδου όταν θα έρθουμε για την επόμενη έκθεση, θα δείτε ότι έχουμε περισσότερες πληρωμές ε, για τα επόμενα χρόνια και λιγότερες δεσμεύσεις, γιατί ήδη έχουν αναλυφθεί οι δεσμεύσεις και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες ε, δεσμεύσεις και λιγότερες πληρωμές. Αυτός είναι ένας κύκλος που έχουμε κάθε φορά και τον γνωρίζετε κι εσείς, είστε εξοικειωμένοι με αυτόν και ε, άλλωστε το Connecting Europe Facility ε, το ε, εξυμνούν όλοι ακριβώς γιατί έχουμε πολύ ταχύ εφαρμογή, μπορούμε να πληρώσουμε πολύ γρήγορα και υπάρχει πολύ μικρή στέρηση στις πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βεβαίω δεν έχει καμία σχέση με τι δεσμεύσει και τι υποχρεώσει. Ε, κάνει απλώ οικονομικέ συμφωνίε και εδώ έχουμε και τα στοιχεία για το τι ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πού πήγαν τα κονδύλια το 2014 και το 2015. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια κατανομή, την οποία θα πρέπει να σας εξηγήσω εν συντομία. Πάνω από το 50% πήγε στους σιδηροδρόμους. Αν δείτε όμως μόνο τα στοιχεία του Connecting Europe ε, Facility, θα το δείτε και στις ε, εκθέσεις, ήμασταν περίπου στο 70% για τους σιδηροδρόμους. Όταν δείτε λοιπόν το συνολικό στοιχείο, τα οδικά δίκτυα και οι άλλες πτυχές ήταν περισσότερο, ε, υψηλότερα, είχαμε 52% συνολικά, αλλά στο Connecting Europe Facility τα οδικά δίκτυα είναι ε, πολύ χαμηλότερα και εδώ βλέπετε και το δικό δίκτυο στην ε, ε πίτα είναι στο 30%. Είναι σημαντικές αυτές οι πληροφορίες για σας για να μπορέσετε να καταλάβετε φυσικά να διαπιστώσετε ότι είναι συμπληρωματικά τα κονδύλια αλλά και διαφέρουν. Το Connecting Euro Facility δίνει περισσότερα χρήματα στους σιδηροδρόμους, ενώ τα άλλα κονδύλια συνεισφέρουν και στο διευρωπαϊκό δίκτυο για τα οδικά ε, δίκτυα και για τα άλλα τμήματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Um, Στην επόμενη διαφάνεια θα ήθελα να σας εξηγήσω και λίγα περισσότερα πράγματα για το πώς υποβάλλεται η έκθεση και πώς ακριβώς έγινε. Γιατί είναι η πρώτη έκθεση που σας κάνουμε βάσει του κανονισμού των διευρωπαϊκών δικτύων και η συγκέντρωση των στοιχείων δεν ήταν πολύ εύκολη. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν πάντα διαθέσιμες πληροφορίες γιατί υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο εθνικοί, θα μπορούσαν να είναι ιδιώτες, ε, τοπικοί, ενδιαφερόμενοι κλπ. Και δεν ήταν πολύ εύκολη στη συλλογή των στοιχείων και μάλιστα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα καθόλου ε, το 2016. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία του 2014-2015, το 2016, αλλά δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει αυτό, διότι πρέπει τα κράτη-μέλη να συλλέξουν τα στοιχεία ε, και μέχρι να τα συλλέξουν ήμασταν ήδη στις αρχές του 2017 και υπήρχαν ε, και ε, συγκεκριμένοι σύμβουλοι και είχαμε και μια έκθεση για να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση των στοιχείων και με όλα τα στοιχεία που είχαμε από τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, ήταν αδύνατο όμως ε, να γίνουν στα πλαίσια του νησιν Δηλαδή το 2016-2017 θα σας το παρουσιάσουμε το 2019. Αυτό δεν γίνεται γιατί δεν θέλουμε να σας διαθέσουμε τα στοιχεία, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να μας δώσουν τα στοιχεία νωρίτερα. Επίσης, για να το βελτιώσουμε λίγο, ε, το Σεπτέμβριο θα γίνει κάτι επιπλέον για το 2016, ώστε να μπορέσουμε να σας δώσουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Αυτά τα έχουμε στην επόμενη διαφάνεια, γιατί ξέρετε ότι δεν θέλουμε να μη σας ενημερώνουμε και θέλουμε να τις έχουμε εγκαίρωσες πληροφορίες και για σας. Ερχόμαστε τακτικά ε, για τα στοιχεία από τους Ευρωπαίους συντονιστές, τους ακούτε τακτικά εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα μέσω των οποίων σας ενημερώνουμε για την εκτέλεση του προπολογισμού, για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά το διευρωπαϊκό δίκτυο, παραδείγματος χάρη τα φυλάδια τα οποία ε, τυπώνονται για τις προσκλήσεις των προσφορών, Επίσης ε, γίνονται και διασκέψεις. Πολύ, συχνά θα, ε, πολύ σύντομα συγγνώμη, θα έχουμε τη διάσκεψη του ε, Connecting Europe Facility το Σεπτέμβριο στο Τάλι. για να μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν τα στοιχεία για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Δημοσιεύουμε και φυλάδια και σας δίνουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσουμε και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την εφαρμογή του Connecting Europe Facility και επομένως και των διευρωπαϊκών δικτύων ε, σε ένα συγκεκριμένο φυλάδιο, ώστε όταν έρθετε στο Ταλίν ε, να έχετε ήδη εκ των προτέρων δύο εβδομάδες πλήρη ε, όλες τις πληροφορίες των, της εφαρμογής των δύο κανονισμών. Και αυτό φυσικά θα σας διαφωτίσει και για τα όσα θα συζητήσουμε στο Τάλιν που θα είναι και η προετοιμασία των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Και όπως σας είπα, ε, κύριε Αντάλη, ήδη έχουμε δέσμευση στο 95% μας έχει μείνει μόνο ένα 4% λοιπόν για τις μεταφορές ε, στο μέσο του Connecting Europe Facility και πρέπει φυσικά να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και θέλουμε να ζητήσουμε από τα μέλη του Κοινοβουλίου να είναι εκεί στη συζήτηση στο Τάλιν. Θα συμπροεδρεύουμε με τον ε, ε, Εστονό Υπουργό και τον Επίτροπο Μπούλτς και θέλουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά εγκαίρως πριν ληφθούν αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω. Όπως σας είπα θα έρχομαι κάθε δύο χρόνια να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Ε, πρόκειται για πολύ καλά στοιχεία, τα οποία εξηγούν τι δουλειά έχει γίνει, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για την πρόοδό μας κάθε δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci beaucoup, Monsieur Reuters. Alors, oui, ça... Σας ευχαριστούμε πολύ. Η στόχη της Επιτροπής μας είναι να έχουμε κανονικό προϋπολογισμό αυτό που θέλουμε είναι να επενδύουμε σε πολιτικές ευρωπαϊκών μεταφορών που έχουν μελλοντικέ προοπτικές και αποτελεί αυτό πραγματικά αναγκαιότητα για την Ευρώπη. Δείχνουμε και στους πολίτες ότι μας απασχολεί το θέμα της κινητικότητας των πολιτών και παράλληλα τηρούμε τους στόχους και λαμβάνουμε υπόψη και τις οικονομικές παραμέτρους. Θα το υπενθυμίσουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστέ, τον κύριο Βιμ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μάρκους Πίπερ ε, μάλλον δεν κατάλαβα ότι άλλαξε η ημερήσια διάταξη Οπότε θα λάβω εγώ το λόγο στη θέση του, γιατί φαντάζομαι ότι θα ήθελε να κάνει αυτές τις παρατηρήσεις για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καταρχήν, ευχαριστώ την ε, Επιτροπή για αυτή την πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση. Δεν ε, μας έχει μείνει καμία ε, αβεβαιότητα. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Ο κ. μας μίλησε για δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 13,69. Ποια ήταν η κατάσταση πριν και μετά το μηχανισμό CF? γιατί ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε υψηλό δανεισμό, και έδινε δηλαδή υψηλά δάνεια και πριν από το μηχανισμό από τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Θα θέλαμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος ε, των Ευρωπαϊκών Διαφορετικών Ταμείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κάτι το οποίο μας ανησυχεί είναι το θέμα των ε, υποχρεώσεων ε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, γίνονται οι αλλά δεν έχουμε στοιχεία για το τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Δεν είναι σωστό να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να μας δώσουν στοιχεία. Κάτι θα πρέπει να μπορεί να γίνει για να το διορθώσουμε αυτό. και είμαι υπεύθυνο και για την επιτροπολογία σε άλλη επιτροπή και πάντοτε είναι ένα θέμα που συζητάμε με την Επιτροπή. θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο ε, να μας δίνουν στοιχεία τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το Ταλίν, ε, φαντάζομαι ότι θα ε, πάνε όλα κατευχήν. Θα φροντίσουμε το θέμα των μεταφορών να τεθεί ως θέμα προτεραιότητας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήξερα ότι είχαμε ε, ένα ποσό 730 εκατομμυρίων, ε, ενώ τώρα μιλάμε για πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Ήταν αρκετά μεγάλη διαφορά από τα 730 δις. Και αν δούμε και τα στοιχεία μέχρι το 2030, ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω ε, για μια ανησυχία μου ότι έχουμε δηλαδή έλλειψη στοιχείων και θα ήθελα να μας διευκρινίσετε με ποιο τρόπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποιο είδος ε, ε, παθητικής αντίστασης προς το Συμβούλιο και στα κρατημέλη για να βελτιώσουν την κατάσταση των στοιχείων των δεδομένων που έχουμε. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω, αν και ξέρω ότι συνεχίζεται η εργασία, με ποιο τρόπο από εδώ, από το Κοινοβούλιο, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ένα είδος μη τέρμα, ας πούμε, γιατί προετοιμάζουμε το επόμενο, το επόμενο PDP, το προετοιμάζουμε ήδη από τώρα ε, και θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες όπως έγινε και την προηγούμενη φορά μέσω πρόθεσμα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε ένα καλύτερο ε, PDP. Έπειτα, οι συντονιστές μπορούν να βελτιώσουν και την, την, την ποιότητα των στοιχείων ώστε να έχουμε μία πηγή, ακριβώ αυτό που είπε ο κύριος Βαντεκά, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από πλευρά των κρατών μελών όσον αφορά όλες τις περιφέρειες. Θα μπορούσατε επίση να μας δώσετε ένα κατάλογο νομοθετικών ετοιμάτων, νομοθετικών σημείων που εντάσσονται σε αυτό το TNT. Ξέρουμε ας πούμε από τους συντονιστές, από τον κύριο Βήμ, ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη νομοθεσία για να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε ε, τα όσα ε, ε υπάρχουν ως στοιχεία στον δημόσιο τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες. Και πρέπει να δούμε επίσης αν η Κομισιόν μπορεί να μας βοηθήσει να τονίσουμε, να υπογραμμίσουμε την αποτελεσματικότητα όλου αυτού του μέσου ε, σε σχέση με άλλα ε, μέσα που δεν είναι τόσο ικανοποιητικά και τόσο αποτελεσματικά. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να το δείξουμε αυτό. Και τέλος, ένα τελευταίο αίτημα, να έχουμε μια τέταρτη στήλη για να δούμε πώς πάνε οι δαπάνες των κρατών για τις υποδομές. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο ε, πέρα από τις δεσμεύσεις υπάρχουν και, υπάρχει και δράση. Ευχαριστώ. Α, κυρία Φώστερ, θέλετε το λόγο? Όχι. Οπότε εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλημέρα στον ε, Διευθυντή. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση αυτή. Έχω μια-δύο παρατηρήσεις σε σχέση με τις δύο στήλες πάνω από το 75% και κάτω από το 75%. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε τι ακριβώς σημαίνει κάτω από το 75%. Ε, αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση ε, Είμαι ευτυχής που το ΤΕΝΤΗ και το ΣΕΦ είναι επιτυχή όσον αφορά την, την ε, δέσμευση των ε, κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ φρόστεκτο, αλλά έχω την εντύπωση ότι κοιτάζουμε περισσότερο τις λεπτομέρειες εδώ ε, και μόνο από οικονομικής άποψης. Λες και είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμού. Δεν λέω ότι απαραίτητο τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά θα ήταν ίσω καλός για την επόμενη παρουσίαση να εξετάσουμε και τι διαφορά έχει κάνει αυτό σε σχέση με τις πραγματικές μεταφορές. Πέρα από τις μελέτες σκοπιμότητας σε σχέση με το TNT και τα λοιπά που δείξαν ότι θα πρέπει αυτό να οδηγήσει σε ε, καλύτερες ροές εμπορίου, καλύτερη ροή της κυκλοφορίας κτλ. Δεν, δεν, δεν αναζητώ δηλαδή κάποια τεράστια μελέτη, αλλά θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ε, για να δούμε αν όντως οι μελέτες σκοπιμότητας έδειξαν ε, σωστά ε, ότι έπρεπε να γίνει το α ή το β και να χρηματοδοτηθεί. Και αυτό να το δείξουμε, μπορούμε να το δείξουμε και τόσο σε εμπειρογνώμονες όσο και σε μη εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω αν θα είμαστε στο πρώτο ήμιση, στο δεύτερο ήμιση, αν θα είμαστε ακόμα εδώ ή όχι, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε από την άποψη της απόδοσης το πράγμα. 2% για τις πολυτροπικές, εγώ δεν είμαι ειδικό, αλλά και πάλι για μένα ε, σημαίνει ότι αυτό θα είναι πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Και όσον αφορά τα στοιχεία, Ξέρω πως η Κομισιόν είναι σε δύσκολη θέση, αλλά αυτό με φέρνει και πάλι στις διάφορες τακτικές εκθέσεις και αναφορές στο παρελθόν, ιδιαίτερα για, τις, για τα μη μέλη. Τη στιγμή δηλαδή που κάτι καθίσταται ορατό, αυτό επιβάλλει μεγαλύτερη πίεση Εγώ ως ε, πρόεδρος θα ήμουν πολύ ε, δύσκολη θέση αν ε, κάποια θέση είναι κενή ενώ οι Ισπανοί ας πούμε το συμπληρώνουν πάνω από 25%. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε αυτά τα στοιχεία, δεν χρειάζεται απόφαση εδώ. Είναι μια ένα πολιτικό αίτημα που υποβάλλουμε. Ε, Επίση στο μέλλον, ξέρω πως ε, τα, τα έχουμε από του συντονιστέ, την αξιολόγηση της πρόοδου στα διάφορα ε, τμήματα του TNT. Αλλά θα ήταν καλό την επόμενη φορά να δούμε μια αξιολόγηση του πώς προχωράει το ΤΕΝΤΗ, όχι με βάση το πόσο έχουμε χαλάσει, αλλά το όσον αφορά την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Γιατί αυτό δείχνει πώς θα πάνε τα κράτη, αλλά και πώς θα πάνε οι συντονιστές. Ξέρω πως γενικά είναι καλά τα αποτελέσματα. Αλλά... θα πρέπει να το δούμε. δεν θέλω να είμαι αγενής στους συναδέλφους, γιατί και εγώ είμαι συντονιστής, αλλά πρέπει να δούμε τη γενική εικόνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τελίντσα. Έχω και εγώ πολλές ερωτήσεις. Πρώτη είναι, η Κομισιόν έχει ήδη ένα νέο νομικό πλαίσιο, ένα νέο project. Γιατί αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα χρειαστούμε ένα νέο νομικό πλαίσιο. Και εφόσον θέλουμε κάτι τέτοιο να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί ο επόμενο προπολογισμό θα φτάσει επίση πολύ γρήγορα. Η επόμενη μου ερώτηση είναι πολύ απλή και θα σα ε, ενοχλήσω με εκείνο το ε, Λιόν Τωρίνο, αλλά εγώ διαπιστώνω πως η, κυβέρνησή μου λέει ίσως πρέπει να σταματήσουμε τέτοια project. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς τεχνικά μια κυβέρνηση, όποια και είναι η χώρα, σταματά ένα μεγάλο έργο. Τι θα γίνει. Παίρνει πίσω τα λεφτά η Κομισιόν. Να μου εξηγήσετε πώς γίνεται. Έχει... Α, όχι. Έχει και... Έχουμε και τον κύριο Έρτου που ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόιτες για την παρουσίαση αυτή. Πάντα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τις θετικές εξελίξεις και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και ο συνάδελφος Ταλίτσκα, ήθελα και εγώ να πω ότι στην Επιτροπή Μεταφορών είχαμε μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση που χρειαζόμαστε από τα κράτη-μέλη. Τονίζω για άλλη μια φορά την ανάγκη να έχουμε τέτοια στοιχεία. Εποφελούνται τα κράτη-μέλη από τη χρηματοδότηση και χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να μπορούμε να προγραμματίσουμε και την μελλοντική μας πολιτική. Υποστηρίζω και εγώ λοιπόν την πρόταση αυτή. Και έχω μια σύντομη ερώτηση. Έχουν ήδη δαπανηθεί το 90% του προϋπολογισμού ε, και το κύριο σημείο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Γνωρίζουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών πολύ καλά. Οι προτάσεις είχαν γίνει τα τελευταία, πριν από πέντε χρόνια και τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά όσον αφορά την κινητικότητα. Αυτό που είχαμε κατά νου είναι ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε αυτό το πακέτο και μετά μια νέα πολιτική και νέα μέτρα μέχρι το 2030. Το δεύτερο μέρος των όσων είχαμε κατά νου να κάνουμε ίσως πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά. Δηλαδή, το μέλλον των μεταφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όταν λέω το μέλλον των μεταφορών, έχω κατά νου μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αλλά πολλές χώρες, ε, όπως ε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, οι κινητήρες δίζελ, ε, οι τεχνολογίες και η εξέλιξή τους ε, και εδώ και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι πολλές οι εξελίξεις και όλες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ε, σε αυτή τη συζήτηση ποια είναι η κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε για την κινητικότητα στην Ευρώπη. Μπορούμε να υποφεληθούμε Τη ε, ευκαιρία ε, για την οδηγία για την έγκριση τύπου ή για τα ε, οξύδια του αζότου. Έχουμε ευκαιρίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπούμε στη συζήτηση αυτή και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν της περίοδου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ίσως θα πρέπει να διαμορφωθεί με έναν άλλο τρόπο. Δεν μιλάω για ένα master plan αλλά ένα μεγάλο σχέδιο που θα δίνει την κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10, 15, 20 χρόνια. Όταν μιλάμε για ε, ηλεκτρισμό και κινητικότητα και τεχνολογία υδρογόνου, η βιομηχανία μας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση γιατί έχουν μια προοπτική 5-7 χρόνων και δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο στην Ευρώπη, ούτε μπορούμε να το κάνουμε μόνο στη Γερμανία. Πρέπει να ξέρουμε στην αλυσίδα παραγωγής τι ποσοστά ε, προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια, τι μπορούμε να προβλέψουμε για τα επόμενα 20 χρόνια, για να επιτύχουμε τους στόχους μας σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά και το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ρετούκ. Τα ερωτήματά σας είναι συναρπαστικά, κύριε Ερτουκ. Δεν με ακούτε. Ναι, σε εσά μιλούσα, αλλά δεν είχατε ακουστικά. Έλεγα, κύριε Έρτουγκ, ότι είναι κλειδί η ερωτήση για το μέλλον. Όσον αφορά τη μεταστροφή της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας, πώς θα συνοδεύσουμε αυτή την μετατροπή πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις ε, να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό αυτού του κλάδου. Μιλήσατε για το υδρογόνο, για τον ηλεκτρισμό και εγώ θα προτιμούσα να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι πυρηνική ενέργεια, φυσικό αέριο και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να προβλέψουμε για το μέλλον. Όταν μιλάμε για την αυτοκινητοβιομηχανία, πρέπει να λάβουμε την τεχνολογία υπόψη. Και εσείς κυρία του που ασχολείστε και με τα αυτόνομα οχήματα κλπ. Ξέρετε ότι έχουμε καθυστερήσει και δεν μπορούμε να μιλάμε για μετασχηματισμό του κλάδου αν δεν μιλάμε και για επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Υπενθυμίζω ότι αν δείτε τα στοιχεία στην Ευρώπη για τους υπαλλήλους στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι 15 εκατομμύρια. Η πρόκληση μεγάλη λοιπόν. Συμφωνώ λοιπόν με σας κυρία Τούκ, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια περίοδο μόνο 7 ετών. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι μέσα στις ε, ηγετικές χώρες του κόσμου, γιατί βλέπουμε ότι και η Ιαπωνία και, τα, και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν περάσει σε κάτι άλλο στην αυτοκινητοβιομηχανία και πρέπει και εμείς ε, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ρόιτες για να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Πολύ καλές οι ερωτήσεις σας, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ακούσαμε. Γυρίσατε από διακοπές με ξεκάθαρο μυαλό και με πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις. Για τις ερωτήσεις του κ. Βαντενκάμ πρώτα. Όντω στην έκθεση αυτή για το 2014 και 2015, η διευκόλυνση για την Ευρώπη δεν φαίνεται ε, τόσο έντονα, γιατί ήταν η αρχή της απόφασης να έχουμε την ε, διευκόλυνση για την Ευρώπη είχε βγει με ένα κονδύλι 2,2 δισεκατομμυρίων. Στην επόμενη έκθεση λοιπόν θα δείτε καλύτερα τι έχει γίνει με τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και τον μηχανισμό διευκόλυνση για την Ευρώπη. Τώρα θυμάμαι ένα ποσό 1,4 δισεκατομμύρια για επενδύσεις. Θα το λάβετε στο έγγραφο που θα λάβετε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα αυτό είναι αυτό που θυμάμαι μόνο από μνήμης. Ε, και είναι σημαντικό να δούμε και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των δανείων και τις πλατφόρμες και μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί. δεν το βλέπετε στην έκθεση για το 2014, αλλά θα φαίνεται στην επόμενη έκθεση. Εσείς αναφέρετε και το θέμα των στοιχείων που δίνουν τα κράτη-μέλη. Η υποβολή εκθέσεων ε, γίνεται εξαιρετικά όσον αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της ε, διευκόλυνσης για την Ευρώπη. Γιατί έχουμε άμεσο διάλογο με τα κράτη-μέλη και με τους ε, Υπευθύνου των έργων και έχουμε επακριβή στοιχεία για όλα, τα, για όλα θέματα του προϋπολογισμού, για όλα τα έργα. Ξέρουμε πού πάνε τα κονδύλια και ποιες δράσεις έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όπου έχουμε αποκεντρωμένη διαχείριση, είναι πιο δύσκολο να λαμβάνουμε στοιχεία, γιατί χρειάζονται περισσότερο χρόνο οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο να πάρουν τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Μπορεί λοιπόν η υποβολή εκθέσεων ε, από τα διαφθορτικά ταμεία να γίνεται λίγο, με λίγη καθυστέρηση. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους ε, της Γενικής Διεύθυνσης Ρίτζιο. αλλά για άλλα τμήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μπορεί να έχουμε ε, λιγότερο καλή εικόνα και χρειάζεται περισσότερος χρόνος μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία. Εάν ε, τώρα μιλήσουμε και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ξέρουμε τη χρηματοδότηση που δίνεται και όλα αυτά αποτελούν τμήμα της χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που γνωρίζουμε. Πέραν όμως αυτών που σας παρουσίασα και εγώ στην παρουσίασή μου, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας υποβάλουν εκθέσεις για όλες τις επενδύσεις που κάνουν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά αυτές οι πληροφορίε έρχονται από πολλέ πηγές και από περιφερειακές και από τοπικές αρχές και από ιδιωτικούς φορείς, ε, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Και είναι πιο αργή η ροή πληροφοριών. Αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, και ο κύριος Τελίτσικα το ενέφερε, ε, είναι να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουμε μια βάση δεδομένων περισσότερο διαφανή. Και έχουμε τη βάση δεδομένων TEN-TEC, που έχει και ένα δημόσιο κομμάτι και ένα κομμάτι περιορισμένης πρόσβασης μόνο για εμπειρογνώμονες. Το κομμάτι που είναι ανοιχτό δημόσια μπορείτε ακόμη και από το τηλέφωνό σας να το συμβουλευτείτε και να δείτε διαφανέστατα τα στοιχεία για τις δράσεις των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια λιγότερα στοιχεία για τα άλλα θέματα που ρώτησε και ο κύριος ε, Τελίσκα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και εμείς ξέρουμε ακριβώς το ποσοστό 90-96% ή σε κάποια άλλα 40-50% και θα μπαίνουν και τα κριτήρια σε αυτή τη βάση δεδομένων και θα μπορεί κανείς ε, να μπει στην ενότητα που τον ενδιαφέρει, να δει τα κριτήρια και να δει τα κονδύλια που έχουν ταπανηθεί και από ποιον και όλα τα στοιχεία. Και μέχρι το τέλος του έτους τα κράτη-μέλη περιμένουμε ότι θα επικυρώνουν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων και αφού επικυρωθούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων θα μπορούμε και να τα βγάλουμε δημόσια. Θα έχουμε λοιπόν όλο και περισσότερα στοιχεία διαθέσιμα για το κοινό. Πολύ σωστή η παρατήρηση σας κύριε Τελίσκα ε, και για την επόμενη υποβολή εκθέσεων θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμη καλύτερη παρουσίαση. Θα μπορείτε να δείτε τι έχει χορηγηθεί και τι έχει χρησιμοποιηθεί και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι επενδύσεις με βάση τα διάφορα κριτήρια. Ακόμη για τον προϋπολογισμό, τα, το στοιχείο είναι 750 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να επιβεβαιώσουν αυτόν τον προπολογισμό πριν από τη συνάντηση στο Τάλιν και μα το επιβεβαίωσαν και στα στοιχεία που θα πάρετε την επόμενη εβδομάδα θα δείτε τι προβλέπει κάθε κράτο μέλο να επενδύσει για τις βασικές δράσεις και για το σύνολο των δράσεων και είναι επικυρωμένα τα στοιχεία αυτά. Το 1,53 που αναφέρατε είναι οι βασικές δράσεις και οι ολοκληρωμένες δράσεις και κάποιες ε, επιπλέον δράσεις. Είναι περισσότερο λοιπόν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 1,53. Αυτό που ανέφερε η κυρία Γιάννη Σέντερ για την έλλειψη δεδομένων από τα κράτη-μέλη, το ανέφερα ήδη. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, γιατί και τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιούν το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη. Είναι ένα άμεσο μηχανισμό, του αρέσει αυτή η άμεση διαχείριση. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν τι έχουν να λαμβάνουν Άρα νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη μερικές φορές έχουν δυσκολία να πάρουν στοιχεία από ιδιωτικούς φορείς, όπως είπαμε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ή λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Οι συντονιστές έχουν μια καλύτερη εικόνα γιατί κάνουν τις συναντήσεις με όλους τους εμπλεκομένους και έχουν ε, καλά αναλυτικά δεδομένα. Και τα στοιχεία για τα 750 δισεκατομμύρια, κύριε Βάντεν έρχονται και από τους συντονιστές που έχουν τα λεπτομερή στοιχεία και τη λεπτομερή πληροφόρηση. Στον κύριο Τελίσκα απάντησα ήδη για τα διάφορα μέσα που έχουμε, τη βάση δεδομένων, την υποβολή εκθέσεων κλπ. Για το αν μπορούμε να αξιολογήσουμε την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των διαδρόμων και των συντονιστών. Αυτό ε, είναι κάπως λεπτό σημείο. Και εσείς είστε υπεύθυνο ε, για τη Βόρεια Θάλασσα και την Βαλτική και ξέρετε συντονιστής ότι είναι δύσκολο, γιατί μερικές φορές δουλεύετε σε ένα έργο επί χρόνια, ε, αλλά είναι δύσκολο να έχετε μια τόσο ξεκαθαρή εικόνα. Τα εργαλεία που έχουμε τώρα είναι καλύτερα, γιατί οι συντονιστές έχουν δυνατότητα να χειριστούν τον προϋπολογισμό και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Με την κυρία Τραουτμάν παραδείγματο χάρη, δουλεύουμε πάνω σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο για να μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα και του νομικού πλαισίου για το που δαπανώνται τα χρήματα. Να μην έχουμε μόνο την προσέγγιση της συμφωνίας επιχορήγησης. Και έρχομαι στη δική σας παρατήρηση, κυρία Νταλή, για το τι συμβαίνει όταν έχουμε καθυστέρηση σε κάποιες δράσεις. Από την ε, εμπειρία μας και από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ξέρουμε ότι κάποιες δράσεις καθυστερούν. Και υπάρχει η αρχή του ότι αν δεν χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια, χάνονται. Τα χρήματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο μιας σύμβασης επανέρχονται στο δικό μας προϋπολογισμό και είναι και πάλι διαθέσιμα για άλλες δράσεις οι οποίες ε, προχωρούν με ταχύτερο βήμα. Αν κάποια δράση όπως η σύνδεση στο Τωρίνο δεν υλοποιηθεί παραδείγματο χάρη και αν δεν ε, ε, χρησιμοποιηθεί και κατά τα τρία επιπλέον χρόνια τα οποία προβλέπονται για να ολοκληρωθεί η δράση, Αν παρόλα αυτά δεν έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια για τις προβλεπόμενες δράσεις, επανέρχονται τα χρήματα στον προϋπολογισμό και προκυρήσονται εκ νέου. και νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ αυστηρό τρόπο διαχείρισης και είμαστε πολύ περήφανοι που η διαχείριση για το ΙΝΕΑ γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι πολύ τομή στην Ευρώπη όπου υπάρχει τόσο προσεκτική και αυστηρή διαχείριση. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις και ο προϋπολογισμός μας είναι μικρός, επομένως δεν μπορούμε να χάσουμε καθόλου κονδύλια. Και τέλος επανέρχομαι στο σημαντικό ερώτημα του κυρίου Έρτογκ. Είπατε και εσείς ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και το θεωρείτε και εσείς σημαντικό. Δεν υποτιμούμε το έργο το οποίο έχετε κάνει, γιατί ο κανονισμός ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι τόσο σύγχρονος, που ήδη διαθέτει μεγάλα ε, ποσά για τα εναλλακτικά καύσιμα και τον εξυγχρονισμό δικτύων. Ένα άρθρο άρθρο αφορά την καινοτομία και ένα άρθρο αφορά τα καινοτόμα καύσιμα και τις αστικές μεταφορές. Αυτά δηλαδή υπάρχουν ήδη στην νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από εσά και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα της, ε, των, ε, της δέσμης μέτρων κινητικότητας και το καλοκαίρι συζητήσαμε κάτι και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δέσμες μέτρων και προτείνει μέτρα η Επιτροπή με βάση αυτά που υπήρχαν στην πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Υπάρχει μέτρο για τα εναλλακτικά καύσιμα και τις υποδομές για να αποφύγουμε ε, το φαύλο κύκλο του αν έχουμε αρκετούς ε, σταθμούς ε, επαναφόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων, αν έχουμε υποδομές για να, να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μισό δισεκατομμύριο και υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης περισσότερων κονδυλίων και κατά την τρέχουσα περίοδο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και γι' αυτό και ε, χαίρομαι που τα συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Ρότερς Χέραλτ, αν μου επιτρέπετε να σας φωνά, αποκαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Είναι πάντα χαρά να σας ακούμε και το γεγονός ότι είστε διαθέσιμος για την Επιτροπή μας μας χαροποιεί. Θα τα ξαναπούμε σε 10 μέρες στο Ταλίν. Ως συνήθω θα έχουμε μια καλή ομάδα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να είμαστε φιλόδοξοι και επικοδομητικοί, γιατί αυτό χρειάζεται η πολιτική μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το χρόνο που μας διαθέσατε και να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η ε, τακτική συνεδρίαση εδώ. Πέραν των συντονιστών βεβαίως, 11 και 5 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές εδώ και οι υπόλοιποι θα τα ξαναπούμε στις 7 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε με τους συντονιστές στις 11 και 5. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιτερς για την ε, ποιότητα των ε, ε, παρουσιάσεών σας και των προτάσεών σας.